Good morning, colleagues. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καταρχήν, αν θέλετε να εγκρίνετε την ημερησία διάταξη, έχετε σχόλια, όχι ευχαριστώ. Εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω στις 12 ε, θα κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε το σχέδιο σύστασης μας βάσει του Άρθρο 55 για δεύτερη ανάγνωση σε σχέση με το σημαντικό θέμα της ε, έκπλησης βόμικου χρήματος και μεταφοράς κονδυλίων. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε την ε, κάρτα ψηφοφορία σας για αυτή τη συνεδρίαση. Επίσης για τους ε, τριλόγους που συνεχίζονται. Καταρχήν επεντεύχθη καλά νέα πολιτική συμφωνία στην οδηγία για τις για, για τις πληρωμές. Συγχαίρουμε τον ε, εισηγητή μας και τον αντιπρόεδρο Μάκους Φέρμπερ, ο οποίος προείδρευσε του τρίλογου αυτού. Το Συμβούλιο έχει κάνει σημαντικές κινήσεις προς την κατεύθυνση του Κοινοβουλίου, επομένως το συμβαστικό πακέτο έχει λάβει υπόψη πολλές από τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και τους παρόχους τους τρίτους παρόχους για τις πληρωμές τα θέματα των ε, εργαλείων πληρωμής και η εξαίρεση για τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. Περιλαμβάνεται επίσης τη συμβαστική λύση η ρύθμιση για την ε, εποπτεία, για τις εξορικαστικές λύσεις. Μπορούμε λοιπόν να τονίσουμε ότι υπήρξε σημαντική ε, πρόοδος σε σχέση με θέση του Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο για την εξαίρεση σε ό,τι αφορά τι τηλεπικοινωνιακέ εταιρείε. Υπήρξε η Γενική Συμφωνία για τη δέσμευτη μέτρο και πρέπει να συνεχιστεί η τεχνική επεξεργασία για να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο κείμενο, αλλά έχουμε την πολιτική συμφωνία. Για το πρόγραμμα στρατηγικών επενδύσεων κάναμε, τρεις, κάναμε δύο τριγωνικούς διαλόγους ήδη για το πακέτο Juncker στο Κοινοβούλιο και μετά στο Συμβούλιο. Ο τρίτος ε, τριγωνικός διάλογος θα λάβει χώρα αύριο. Προχωρούμε λοιπόν με γοργά βήματα, Όντα προσιλωμένοι στο να πετύχουμε με το ταχύτερο δυνατό τρόπο μια συμφωνία για να μπορέσει ήδη το καλοκαίρι να εγκριθεί οριστικά το πακέτο αυτό. Έχουμε φυσικά συμφωνήσει για τη μεθοδολογία, έχουμε ορισμένες βασικές αρχές που συμφωνήσαμε για τη διαδικασία. Αλλά δουλεύουμε σκληρά για ορισμένα θέματα όπου αποκλίνουν οι θέση του Συμβουλίου από το Κοινοβούλιο. Η τρίτο θέμα η έκθεση για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ο πρώτος ε, τριγωνικός διάλογος έγινε στις 25 Απριλίου και τα κύρια πολιτικά θέματα Υπάρχει συμφωνία όλων των θεσμικών οργάνων σε σχέση με τους κοινούς στόχους, παραμένουν ακόμα κάποιες διαφορές, αλλά υπάρχει γενικά αισιοδοξία για το θέμα αυτό. Η συνέχεια των διαπραγματεύσεων θα γίνει στις 20 Μαΐου και συνεχίζεται η τεχνική επεξεργασία. Αυτά υπό μορφή ανακοινώσεων. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 της ημέρησης διάταξης. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση για το ευρώ μέσα στα πλαίσια στα πλαίσια των διεθνών ρυθμιστικών φορέων για τα χρηματοπιστωτικά θέματα και τις συναλλαγές. Η κυρία Γκουλάρ είναι η συγήτρια. Και απλώς υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μελετών που είναι στη διάθεσή μας. Έχουν μεγάλη σημασία λοιπόν όλες αυτές οι αναλύσεις και δείχνουν ποιος είναι και ο ρόλος της Κομισιόν σε όλα τα διεθνή φόρα και όλα αυτά που βλέπουμε από τις μελέτες επιβεβαίωσαν την ανάγκη μιας τέτοιας έκθεσης ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η σχέση της Κομισιόν με το Κοινοβούλιο σε αυτούς τους στρατηγικούς χώρους. Σιλβή, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ όσους παρόντες. Καταρχάς για, την, για το πεδίο αυτής της έκθεσης είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση των 28 ουσιαστικά στα πλαίσια ενός οργανισμού. à remercier Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι πράγματι μας έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της γραμματείας όπως επίσης και των υπηρεσιών τεκμηρίωσης που ε, συντόνισαν τις μελέτες αυτές τις οποίες κρίνω πάρα πολύ χρήσιμες. Ε, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης αυτής της έκθεσης. Καταρχάς, να μην ξεχνάμε ότι η διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι μια πραγματικότητα η οποία αναπτύσσεται συνεχώς. Οι, χρηματοπιστωτικές ροές είναι συνεχείς, χωρίς σύνορα και πράγματι υπάρχει ανάγκη όπως και στο περιβάλλον να υπάρξει μια διακυβέρνηση κοινή με κοινού κανόνες, κάτι το οποίο υπογραμμίστηκε πολύ στο τέλος και γι' αυτό εξελίσσεται σιγά σιγά και η ομάδα των 20, των G20 όπως λέμε και στο οποίο θα επανέλθω. Πάντως στόχος ε, ε, αυτής της έκθεσης δεν είναι λοιπόν να αρνηθούμε αυτή την ανάγκη διεθνοποίησης. Πρέπει να συνεργαστούμε με άλλες χώρες. Είπα, Ασία, η οποία παίρνει όλο και πιο μεγάλη θέση και άλλες αναδιόμενες περιοχές στον κόσμο να συνειδητοποιήσουμε το βάρος του φαινομένου αυτού. Δεν θέλουμε εμείς να αναδιπλωθούμε, δεν θέλουμε να αποκλειστούμε. Θέλουμε να δούμε τι αλλαγές μπορούμε να κάνουμε και σαν Ευρώπη πώς μπορούμε να αμυνθούμε. Υπάρχουν δύο θέματα. Βέβαια αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι η πρώτη συζήτηση και γι' αυτό περιμένω να συνεργαστώ με τους σκιώδεις όλων των πολιτικών ομάδων. Ε, είναι το διακύβευμα στρατηγικό, είναι το διακύβευμα μεσοπρόθεσμο, αφορά την προστασία των συμφερόντων μας σε όλο τον κόσμο και ελπίζω να κάνουμε μια δουλειά η οποία θα είναι κυρίως συλλογική. Ήδη όμως διακρίνω δύο θέματα. Πρώτον, θα πρέπει να απαντήσουμε στους πολίτες μας. Στο ερώτημα το απλό. Ποιος αποφασίζει. Οι πιο απλές ερωτήσεις είναι και οι πιο δύσκολες. Τα παιδιά μας μας το μάθανε αυτό. Ποιος παίρνει αποφάσεις στον οικονομικό τομέα. Μέσα σε ένα σύστημα όπου υπάρχουν ε, εκλεγμένοι εκπρόσωποι, υπουργοί, εθνικά κοινοβούλια, ευρωπαϊκές αρχές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξωτερικές υπηρεσίες, αλλά σε ποιο βαθμό υπάρχει μια διαδραστικότητα ανάμεσα σε αυτά τα όργανα ε, και σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς. Υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας εδώ και αυτή η έλλειψη διαφάνειας μπορεί να οδηγήσει σε μια σύγχυση και απώλεια εμπιστοσύνης. Δυστυχώς και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια απώλεια εμπιστοσύνης απέναντι σε αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν. Τεχνοκρατία, πολιτοκρατία, πολλές φορές οι πολιτικοί δεν γνωρίζουν τι κάνουν οι τεχνοκράτες και ε, επίσης ισχύει και το αντίθετο. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσω μελετών παράγονται ορισμένα υποχρεωτικά σε εισαγωγικά υποχρεωτικά επίπεδα που δεν είναι υποχρεωτικά τελικά, είναι προσανατολισμοί. Οι προσανατολισμοί αυτοί είναι όμως διεθνείς, λαμβάνονται σε επίπεδο διεθνές και γι' αυτό επιβάλλονται. Οι διοικήσεις οι εθνικές τις χρησιμοποιούν και το ίδιο κάνουν και οι επιχειρήσεις, αν και δεν πρόκειται για θετικό δίκαιο. Ξέρουμε την Επιτροπή της Βασιλείας, σαν παράδειγμα, τι προσανατολισμούς έχει δώσει για να υπάρξει ένα ισότιμο πεδίο δράσης με τις Ηνωμένε Πολιτείες και με άλλες εθνικές ειδικαιοδοσίες. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις διαφορετικές. Η αγορά χρηματοδοτεί πολύ λιγότερο την οικονομία από ότι οι τράπεζες στην Ευρώπη. Έχουν υπάρξει ορισμένοι προσανατολισμοί πριν από την υιοθέτηση του κειμένου και υπάρχουν επίσης και δηλώσεις μη συμμόρφωσης, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη ε, τις ε, αποφάσεις τις οποίες εμείς έχουμε λάβει. Δεν θα περάσω σε περισσότερες λεπτομέρειες, σήμερα θα μείνουμε σε ένα πολύ γενικό επίπεδο. Υπάρχει όμως μια θεά περιοχή στο εσωτερικό της οποίας δεν ξέρουμε ποιος παίρνει αποφάσεις, ποιος παίρνει δεσμευτικές αποφάσεις ποιος παίρνει αποφάσεις οι οποίες είναι συμβουλευτικές. Υπάρχουν επίσης θέματα νομικά εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις παραδοσιακού τύπου όπως το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, όπως ο ΟΣΑ και υπάρχουν και άλλες οργανώσεις ιδιωτικού δικαίου οργανώσεις οι οποίες ε, δεν έχουν καν νομική ύπαρξη όπως το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ταμείο Σταθερότητας. Υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας λοιπόν. Είμαστε σε μια κοινωνία η οποία δικαιολογημένα ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια, πρόσβαση σε έγγραφα, πρόσβαση σε πρακτικά συνεδριάσεων. Ο κόσμος θέλει να γνωρίζει τις θέσεις των μεν και των δε. Η διαφάνεια είναι μία από τις κόκκινες γραμμές αυτής της έκθεσης. Εμείς δεν θέλουμε να παρέμβουμε στο πεδίο των εμπειρογνωμόνων. Δεν θέλουμε να μειώσουμε τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων, αλλά θέλουμε σε πολιτικό επίπεδο να γνωρίζουμε τι γίνεται, πώς γίνεται και ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Και τέλος η διαφάνεια αυτή θα επιτρέψει επίσης να μιλήσουμε και για το accountability. Ποιος είναι εμπασπέτος υπόλογος απέναντι στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, και εδώ έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν στον χρηματοπιστωτικό τομέα τρομακτικά λάθη. Ένας από τους λόγους που βιώσαμε τις προηγούμενες κρίσεις είναι ότι οι εμπλεκόμενοι που ήταν υποτίθεται επιβλεπόμενοι δεν ήταν τελικά επιβλεπόμενοι και ε, ουσιαστικά διέτρεξαν κινδύνους απαράδεκτους. Και τελικά τους έσωσε ε, η αλληλεγγύη των φορολογουμένων, κάτι το οποίο είναι αρκετά περίεργο. Οι μελέτες λοιπόν, οι μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας μας δίνουν ένα πρώτο πανόραμα χρήσιμο. Περιγράφουμε δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται όλοι όσοι εμπλέκονται στον χώρο αυτό, δηλαδή τράπεζες, πιστοτικά ιδρύματα, διεθνείς οργανώσεις. Αυτό είναι το πανόραμα, το περιγραφικό κομμάτι που θα πρέπει να το παρουσιάσουμε με αντικειμενικό τρόπο χωρίς να μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή διαφάνεια και accountability, ποιοι είναι οι υπόλογοι. Ένα δεύτερο θέμα τώρα είναι η προστασία των κοινωνικών συμφερόντων. Με ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται σε όλα αυτά τα, τα... Ε, τα όργανα και ποιος είναι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, ποιες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στις εκτελεστικές αρχές και στις αρχές τεχνικού επίπεδου. Αν πάρετε κάποια παραδείγματα, βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοδεύει ή συνοδεύεται από ε, τα κράτη-μέλη, είναι έξι όπως το Stability Board, είναι νέα όπως το Συμβούλιο της Βασιλείας, Υπάρχει μια σύγχυση, εκπροσωπούμεθα σε επίπεδο ευρωομάδα, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε οργανώσεις όπως ΕΣΜΑ, EBA ή και τις κεντρικές τράπεζες. Γενικά δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς ε, γίνεται σε κάθε όργανο, επειδή και οι ιστορικές καταβολές του κάθε οργάνου είναι διαφορετικές. Δεν θέλουμε να τα εναρμονίσουμε όλα, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο προσπίζεται κανείς το ευρωπαϊκό συμφέρον. Να δούμε αν υπάρχει συμφέρον να υπάρξει μια εκπροσώπηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε λόγω και του μεγέθους και της πολυδιάσπασής μας να επηρεάσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι η λεγόμενη κακοφωνία η Ευρώπη δηλαδή να εκφράζεται με τρόπο άτακτο, οι μεν να μην γνωρίζουν τι λένε οι δε. Και δεύτερον υπάρχει το θέμα των συμφερόντων της Ευρωζώνης. Εδώ βλέπουμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σημαντικότατος ρόλος και σαν κεντρική τράπεζα για το νομισματικό κομμάτι, αλλά και με το SSM για θέματα σταθερότητας. Θυμίζω ότι η έκθεση Λαγοζιέρ στην οποία βασιστήκαμε εμείς για να δημιουργήσουμε τις αρχές εποπτείας ε, υπογραμμίζει τα θέματα αυτά. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθούμε να δούμε με τους υπόλοιπους συνομιλητές που βρισκόμαστε. Οι σχέσεις τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές, να κρατήσουμε δομές ιδιαίτερα ευέλικτες. Άλλοι πιστεύουν ότι απαιτείται μια ισχυρότερη διεθνής οργάνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γιατί όχι όλα να τα εξετάσουμε, να επιλέξουμε και να καθορίσουμε προτεραιότητες. Τερματίζω. Η προσπάθειά μας πρέπει να είναι παιδαγωγική αλλά κυρίαρχα πολιτική πρέπει να εμφυσίσουμε περισσότερη δημοκρατία και accountability μέσα σε ένα τοπίο το οποίο είναι πολύ διασπασμένο και πολυπίκυλο. Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει αναλάβει την υποχρέωση να κάνει προτάσεις επί τη βάση του άρθρου 138 της Συνθήκης για μια πιο ενιαία εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ στα διεθνή όργανα εμείς εντάσσουμε την απόφαση αυτή και στα πλαίσια της μελλοντική μας πολιτικής. Θα συνεργαστώ με τους σκιώδεις και ελπίζω να πάμε καλά. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να ακούσουμε και τους ε, σκιώδεις. Να ακούσουμε την κυρία Πιτικάινεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την κυρία Κουλά που ως εισηγήτρια βάλει την πρωτοβουλία να υπάρξει αυτή η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Γιατί όντως ε, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε πιο λεπτομερώς. Σε γενικές γραμμές να πω ότι συμφωνούμε με όλα τα θέματα που θέσατε προς μελέτη. Να υπογραμμίζω κάποια από τα στοιχεία που θίξατε, όπου έχω την αίσθηση ότι έχουμε κοινά συμφέροντα. Οι χρηματοπιστωτικές ε, αγορές φυσικά και η οικονομία είναι παγκόσμια, αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά τα συστήματα, για οι δράσεις μας βασίζονται σε εθνικά συστήματα, μη σας πω και σε περιφερειακές προσεγγίσεις. Αυτό αφανώς. Κάτι άλλο τώρα που σχετίζεται πάρα πολύ με τα θέματα αυτά. Στην οικονομία μας και στις σχετικές ε, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές. Αντιδρούμε πάντα στην καλύτερη περίπτωση. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε proactivity, δεν μπορούμε από πριν να δώσουμε τα σωστά κίνητρα στα συστήματά μας προκειμένου να σταθεροποιήσουμε τις ε, διακυμάνσεις που είναι αναπόφεκτες και ούτε είναι και κακές απαραίτητα αλλά εν περιπτώσει το εύρος των διακυμάνσεων των κινδύνων των αγορών, των διαφορών στις οικονομίες και των διαφορών ε, στα συμφέροντα. Υπάρχουν λοιπόν τρία θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε με πιο συνεκτικό τρόπο στο μέλλον. Πρώτον, και εδώ παίζει ρόλο αυτή η δημοκρατία που Το θέμα της πολιτικής κατεύθυνσης. Αντιδρούμε πάντα με κατακαιρματισμένες πρωτοβουλίε, νομοθεσίες, με αντιδράσεις σε βάση των κινδύνων και των κρίσεων ε, που μαστίζουν την αγορά ή υπάρχει κάποια προετοιμασία, υπάρχει κάποιος σεβασμός προς τους υπαλλήλους, προς ε, τους εμπειρογνώμονες. σε ό,τι αφορά τη Βασιλεία 3 και 4. Θα μπορούσαμε να δώσουμε την πολιτική κατεύθυνση, την πολιτική ορμή στην ε, πρώιμη φάση της ε, διαδικασίας, όχι τις λεπτομέρειες, αλλά να δώσουμε τα γενικότερα κίνητρα, την κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να κινηθούμε. Δεύτερο θέμα, Και αυτό το βλέπουμε στο πάκο των εγγράφων που έχουμε. Ευχαριστούμε τη γραμματεία που προετοίμασε τις μελέτες αυτές. Ο αριθμός των θεσμικών οργάνων και η συνεκτικότητα. Η συνεκτικότητα των οργάνων αυτών σε διεθνές επίπεδο. Αυτό αποτελεί την πρόκληση. Η ευρωπαϊκή πολιτική στα θεσμικά όργανα αυτά έχουμε κάποιο ρόλο να παίξουμε. Έχουμε κάποιο μήνυμα που θέλουμε να αποστείλουμε μακροπρόθεσμα και το παρουσιάζουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Και μάλιστα εγκαίρως σε όλες αυτές τις προπαρασκευαστικές δράσεις, σε όλες αυτές τις διεθνείς οργανώσεις. Είμαστε αυτοί που προωθούμε τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των διεθνών οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε μια καλύτερη γενικότερη οργάνωση. Υπάρχει το G20 αλλά έχει διαφορετικές ε, αρμοδιότητες για τις διεθνείς οικονομικές πρωτοβουλίες Αυτό όχι για να υπαγορεύσουμε στι οργανώσει τι να κάνουν, αλλά για να διασφαλίσουμε καλύτερη συνεργασία. Ένα πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι το εξή. Είναι ένα πρώτο καλό βήμα αυτή η προετοιμασία που κάναμε, η μελέτη που κάναμε στην Επιτροπή. Αλλά έχουμε ήδη διάφορα scoreboards για τις εσωτερικές αγορές, για τις διάφορες δράσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν υπάρχει λοιπόν ένας τέτοιο πίνακας, ένα scoreboard για τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το τι συμβαίνει, ποιε ήταν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, ποιος ο αντίκτυπός τους, ποια θεωρούμε ότι είναι τα επόμενα βήματα, οι επόμενες προκλήσεις. Και τα θέματα επί των οποίων θέλουμε να εργαστούμε. Η προάσπιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να δείξω. What is the parliament's right role? Ποιος είναι ο σωστός ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο να μην καθυστερήσουμε και να μην επισέλθουμε σε μεγάλο επίπεδο λεπτομερία, αλλά σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ ε, καταστηντήριες γραμμέ, πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε με σαφήνεια, αλλά και με ευφυα το ρόλο του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή Οίκων σε ό,τι αφορά τη μόνιμη, το μόνιμο ρόλο αντίδραση σε ό,τι αφορά το scoreboard, σε ό,τι αφορά τα διεθνή χρηματοπιστωτικά και οικονομικά ιδρύματα. Ποια είναι η πολιτική μας και πόσο συχνά την προωθούμε. Κάθε χρόνο, μία φορά κάθε θητεία, δύο φορές κάθε θητεία. Ποια είναι η σωστή συχνότητα και ποιος ο συχνός μηχανισμός. Και πώς συμπεριλαμβάνεται ε, αυτό το σχέδιο και αυτή η πολιτική στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Χωρίς να δημιουργούνται ασφαλώς επιπλέον επιβαρύνσεις γραφειοκρατικής φύσεως. Προσβλέπω στην πολύ καλή συνεργασία και πιστεύω ότι έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα. Πολλά μπορούμε να αποκομίσουμε μόνο αν συνεργαστούμε από κοινού. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι και πολύ σημαντικό θέμα. Το μόνο μου θέμα, και θα θέλω να το σκεφτεί η συγγεντρία, είναι ότι ενώ αυτές οι καλές μελέτες ε, καθυστέρησαν. Δεν ξέρω αν είμαι τεμπέλα ή αν άργησα να το διαβάσω. Δεν είχα χρόνο να μελετήσω σε βάθος όλα αυτά τα έγγραφα. Αυτό να ληφθεί υπόψη στο δικό μας χρονοδιάγραμμα. Και να έχουμε πιο πολύ χρόνο για την ε, εργασία μας αυτή. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην πολύ καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ashley Fox. Λάθο, λάθο, Λάθος, λάθος, ντρέπομαι. Η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ παρόλα αυτά, λέει η κυρία Ντελβό. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς την Κουλάρ γιατί πήρε την πρωτοβουλία για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και αυτούς που υπέβαλαν τα κείμενα, τους συγγραφείς των εγγράφων που είναι χρήσιμα, ψαγμένα, τεκμηριωμένα. Λοιπόν, δύο διαπιστώσεις και τρεις ερωτήσεις. Οι διαπιστώσεις είναι προφανείς αλλά πρέπει να τις τιμήσουμε. Ιδιαίτερα αν θέλουν οι εκλογείς μας και το κοινό μας να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο διακυβερνάτε το χρηματοπιστωτικό στερέωμα και ποιοι ασχολούνται εν πάση περιπτώσει με την χρηματοπιστωτική δραστηριότητα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Όλοι συνειδητοποιούμε καταρχάς την αλληλοεξάρτηση των συστημάτων μας και βασικός στόχος είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη δημοσιονομική σταθερότητα. Δεύτερη διαπίστωση είναι η ποικιλία που παίρνουν αυτά τα φόρουμ, η ποικιλία που παίρνουν αυτά τα όργανα, αυτοί οι θεσμοί και ο τρόπος με τον οποίο αλληλοεπιδρούν. Και επίσης και η ποικιλία με την οποία εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικές φορές είναι όλα τα κράτη-μέλη, άλλες φορές είναι κάποια λιγότερα συνήθως τα ίδια. Πολλές φορές ένα θεσμικό όργανο εκπροσωπείται, μερικές φορές εκπροσωπούνται δύο, μερικές φορές οι αρμοδιότητες ποικίλουν, υπάρχει διαφορετική γεωμετρία παρέμβασης και αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην πω ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι ιδιαιτέρως περιορισμένη. Πρώτη ερώτηση, την οποία θα πρέπει να θέσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει αυτά τα διεθνή φόρα. Από ό,τι φαίνεται η αριθμητική, η ποσοτική παρέμβαση δηλαδή είναι ιδιαίτερο υψηλού επίπεδου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα. Εάν οι θέσεις είναι συγκλίνουσες και συνεκτικές, αυτό είναι πλεονέκτημα. Εάν όμως οι εταίροι βασίζονται στην έκφραση των προσωπικών τους ατομικών εθνικών θέσεων, όχι. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η υπεραντιπροσωπευτικότητα των κρατών μελών έχει ήδη τεθεί σε αμφισβήτηση και θα ενισχυθεί αυτή η στάση γιατί πιέζουν και οι υπόλοιπες πλευρές, ε, ε, τα υπόλοιπα τμήματα του κόσμου αυτού και καλό θα είναι να μπορέσουμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Το δεύτερο ερώτημα, εάν η επιρροή κοινοτική είναι αποτελεσματική, αν καταφέρνουμε να κάνουμε τις θέσεις μας να ακούγονται ή μήπω απλά υφιστάμεθα τις θέσεις όλων των υπολείπων. Εδώ νομίζω ότι αν θέλουμε πράγματι να επηρεάσουμε με σημαντικό και θετικό τρόπο απαιτείται μια, ένα συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη πριν από την έναρξη των συζητήσεων. Δεν γίνεται πάντα αυτό, δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η μορφή του συντονισμού καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη γιατί σε πάρα πολλά θεσμικά όργανα η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται από εξωτερικές υπηρεσίες και από θεσμούς με ανεξαρτησία σχετική που δεν δεσμεύονται δηλαδή και δεν συνδέονται ε, με την ε, εξειδικευμένη πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό καμιά φορά είναι και θετικό, συνήθως είναι αρνητικό. Και τρίτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το πώς ασκείται η συγκεκριμένη αυτή επίρροη. Εδώ επανέρχομαι στα θέματα τα οποία έχουν ε, ήδη τεθεί. Τι συμβαίνει δηλαδή με το θέμα της διαφάνειας, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, μπορούμε άραγε σε επίπεδο πολιτικών οργάνων να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, να είμαστε κοντά στις εξελίξεις και ε, το άλλο ερώτημα είναι το της δημοκρατικής νομιμότητας. Εάν οι αποφάσεις, εάν θέλουμε εν πάση περιπτώσει οι αποφάσεις αυτές να γίνουν δεκτές, η αποδοχή έχει σημασία βέβαια, οι πολιτικοί από μόνοι τους δεν μπορούν πια να αποφασίζουν, αλλά αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την αποδοχή των συγκεκριμένων θέσεων απαιτείται μεγαλύτερη και υψηλότερη δημοκρατική συμμετοχή. Και να προσθέσω μια δευτερεύουσα ερώτηση εδώ, το της εφαρμογής. Τι κάνουμε με όλες αυτές τις συστάσεις, με όλες αυτές τις αποφάσεις, πώς τις μεταφέρουμε τις αποφάσεις αυτές σε επίπεδο κοινοτικό είναι κάτι το οποίο γίνεται με χρήσιμο τρόπο, με ωφέλιμο τρόπο. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία τίθενται. Ε, η τεκμηρίωση η οποία μας έχει δοθεί είναι πληρέστατη, πηγαίνει σε βάθος και θέλουμε χρόνο για να τη μελετήσουμε. Εγώ είμαι διαθέσιμη απολύτως προς την κυρία Γκουλάρ να δουλέψουμε σωστά και να βοηθήσουμε στη σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ ο Ashley Fox. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω την Σιλβία και τους άλλους ε, ομιλητές για τη συμβολή τους στη συζήτηση αυτή. Θέλω επίση να ευχαριστήσω τους συντάκτες των ε, εννέα εγγράφων ενημέρωσης που έχουν ε, προσφερθεί για τη συζήτηση. Δεν τα έχω διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια ζήτησα από τους βοηθούς μου να τα διαβάσουμε, Αλλά νομίζω ότι δίνουν μια πολύ καλή επισκόψη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε ένα από τους διεθνείς αυτούς φορείς. Και αυτό το οποίο υπογραμμίζουμε είναι ότι σε κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφορετικό ρόλο αλλά και διαφορετική θέση. Επομένω, το να έχουμε ένα τελείο που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα συμπεράσματα αυτών των εγγράφων θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Με μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι η Σιλβή θα ακολουθήσει μια πραγματιστική και όχι ιδεολογική αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά. Στις παγκόσμιες αυτές αγορές έχουμε πολλούς διεθνείς φορείς που αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς τρόπους και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθήσει διαφορετικούς ρόλους σε αυτούς τους φορείς. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως οι εκλογείς μας ποιος είναι αρμόδιος για να παίρνει ποιες αποφάσεις για τη ρύθμιση των παγκοσμίων αγορών και να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας. Εδώ να προειδοποιήσω είπε η Σιλβία ότι δεν θα πάρει ιδεολογική προσέγγιση. Το χαιρετίζω αυτό. Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση δεν θα γίνει όχημα για να πούμε ότι σε κάθε ένα από αυτούς τους φορείς θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο ρόλος της Ευρωζώνης αντίστοιχα. Κατά την άποψή μου, ο ρόλος του κράτους, έθνους είναι ο χώρος όπου ευδοκιμεί η λογοδοσία. Εκεί λογοδοτούν οι κυβερνώντες. Πολύ σπάνια έρχονται σε μένα οι εκλογείς μου και μου λένε τι κάνετε για να ρυθμίσετε τις παγκόσμιες χρηματαγορές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν και να συντονίσουμε καλύτερα την προσέγγιση μας, όταν λέω εμείς εννοώ τα κράτη-μέλη, πριν από διεθνείς ε, συναντήσεις, αυτό είναι πολύ λογικό, το να προσπαθήσουμε όμως να συντονίσουμε τις προσεγγίσεις μας δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να έχουμε πάντα μια κοινή αντιμετώπιση. Γι' αυτό προσβλέπω στη συνεργασία με την Σιλβή και τους άλλους σκιώδεις και ελπίζω ότι όλοι θα πάρουμε μια πραγματιστική θέση και όχι μια ιδεολογική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Δεν βλέπω τον Γκέλ Όχι. Ο Σβέν Γκίγκολτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και από την δική μας ομάδα θέλω να ευχαριστήσω την Σιλβί Γκουλάρ για την πρωτοβουλία της να επεξεργαστεί το θέμα αυτό. Ήδη οι προτάσεις αυτές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα εργασίας τα οποία παρουσιάστηκαν και τα σχόλια τους δείχνουν ότι εδώ έχουμε ένα κοινό θέμα μια κοινή ανησυχία μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών αρχών. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ήδη λεχθέντα, αλλά Ashley πρώτα απ' όλα. Όλα αυτά που λες δείχνουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να αποχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κανένας άλλος πολιτικός δεν θα παραδεχόταν ποτέ ότι δεν έχει διαβάσει αυτά τα έγγραφα πληροφόρηση και τα αφήνει για τους βοηθούς του. Αυτό δείχνει ότι είσαστε και ανθρώπινοι. Εγώ δεν τα έχω διαβάσει όλα, αλλά η πρόθεσή μου είναι να τα διαβάσω όλα. Αυτό δείχνει όμως γιατί δεν μπορούμε να χάσουμε το βρετανικό φλέγμα και χιούμορ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και αν δεν συμμερίζομαι σου για το κράτος μέλος το εθνικό κράτος ως το ιερό δισκοπότηρο της δημοκρατίας μέχρι το τέλος της ιστορίας. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο ερώτημα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη δική μας πολιτική ομάδα. Δεν είναι τόσο πολύ το πώς θα μεγιστοποιήσουμε την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι θετική αυτή η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συμφωνώ ότι εδώ μπορούμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα για τα πολλά κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται σε αυτούς τους διεθνείς χώρους ενώ άλλα κράτη-μέλη δεν εκπροσωπούνται καθόλου και αν είναι συνολικά δίκαιο να έχουμε τόσο πολλούς Ευρωπαίους εκπροσώπους οι οποίοι απλώς διαφωνούν μεταξύ τους και δεν ασκούν καμία επιρροή στους άλλους και επομένως είναι ασαφής και ο ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν αποδέχονται όλα τα κρατη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να είναι η φωνή της Ευρώπης σε αυτούς τους διεθνείς χώρους. Παραμένουν λοιπόν όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά. Το μεγάλο όμως ερώτημα για μένα είναι είναι αν δεχόμαστε την αρχική ιδέα της Ευρώπης που ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια να, να συμβιβαστεί, να συνενωθεί μάλλον με τη δημοκρατία η μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση. Και έχουμε αναπτύξει για πρώτη φορά κάποια πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας και αχαιρεότητας. Αυτά προσπαθούμε να επιτύχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγχρόνως ξεπερνώντας τα στενά όρια των εθνικών δημοκρατιών. Θα χρειαστούμε περισσότερους χώρους διαφάνειας και λογοδοσίας σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό υπάρχει αυτή η, ανάγκη που οδήγησε σε ένα διεθνές στερέωμα διεθνών φορέων. Τα θέματα λοιπόν αυτά της διαφάνειας, της ε, και της λογοδοσίας θα πρέπει να τεθούν σε όλους αυτούς τους διεθνείς φορείς τα έγγραφα εργασίας καταδεικνύουν ότι αυτό δεν έχει επιτευχθεί στο ίδιο επίπεδο σε όλους τους φορείς. Παραμένουν θέματα όπως ποιος κρατάει την α ή τη β θέση. Είναι θέμα διαφάνειας, ώστε να μπορεί κανείς να γνωρίζει τις θέσεις των, κυ... κυβερνήσεων. Αλλά γνωρίζουμε ποια λόμπι έχουν προσπαθήσει να επηρεάσουν τη θέση των κυβερνήσεων. Ποια είναι τα λόμπι τα οποία λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο και εδώ είναι φανερό ότι η μονομέρεια που βλέπουμε και στις Βρυξέλλες ότι είναι πολύ πιο εύκολο για μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τις ενώσεις ε, πολιτών που νοιάζονται για το κοινό καλό αλλά δεν έχουν απαραίτητη οργάνωση, αυτές οι ανισομέρειες αντανακλώνται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή της ε, Βασιλείας. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια θέματα επιρροής που πρέπει να ληφθούν υπόψη και το ερώτημα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε την διαφάνεια, την ε, ακεραιότητα και τη λογοδοσία όταν πρόκειται για περαιτέρω φορείς όπως ε, αυτούς τους φορείς οι οποίοι θέλουν να δημιουργηθούν στα πλαίσια αυτή τη TTIP. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι ακριβώς επίκαιρη και θα πρέπει να συζητήσουμε και ποιε είναι οι δικέ μα δομέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ποιο τρόπο εξασφαλίζουμε την ε, λογοδοσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώ εξασφαλίζουμε ότι είναι υπόλογοι για τη δράση τη μέσα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ μπορούμε να θέσουμε ερωτήματα για τα θέματα αυτά, αλλά δεν τα ρωτάμε πάντα, δεν τα θέτουμε αυτά τα ερωτήματα πάντα. Θα πρέπει λοιπόν να αυτοερωτηθούμε για το κατά πόσο η δημοκρατική διαδικασία που θεσπίζεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας περιορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σε διεθνείς φορείς είτε στην ε, λειτουργία την, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στην επιρροή που ασκεί. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω περισσότερα για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ε, κύριε Μπερές. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συζήτηση την οποία ξεκινάμε είναι σημαντική. Στα πλαίσια της συζήτησης αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέμβει περισσότερο από ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγα. Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο διαστάσεις οι οποίες μου φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Η πρώτη αφορά το θέμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς δηλαδή όταν εκφράζουμε τις θέσεις μας σε εξωτερικό επίπεδο όπου υπάρχουν αρμοδιότητες εθνικές παρόλα αυτά τα κοινοτικά όργανα μπορεί να λειτουργούν σαν εκφραστές οι λογιστικοί κανόνες, σαν παράδειγμα. Έχουμε την έκθεση της ΕΦΡΑΓ, όπου λέγεται ότι στην αρχή είχαμε εφεύρει, αν θέλετε, αυτούς τους κανόνες, για να εκπροσωπείται σωστά μέσω της ΕΦΡΑΓ Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα πράγματα λίγο εδώ σε εισαγωγικά τούμπαραν. Η Στατιστική Υπηρεσία ε, παρουσίασε μια πρόταση η οποία οδήγησε σε κάποιες αλλαγές αλλά τελικά σε επίπεδο λογιστικών κανόνων το θέμα δεν είναι να μεταφέρουμε τους διεθνείς κανόνες σε μας, αλλά το να συντονίσουμε το τι κάνουν τα, οι εθνικές αρχές. Οπότε τίθεται εδώ σαφώς το θέμα της ε, επικουρικότητας. Και αυτό επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα κοινοτικά συμφέροντα. Αυτή ήταν μια πρώτη ανησυχία επιμέρους. Η δεύτερη τώρα Έχουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες αναλάβει οι οποίες είναι διαφορετικού χαρακτήρα μεταξύ τους. Εδώ τίθεται ξανά το θέμα της ε, αντιπροσώπευσης των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο σε επίπεδο βασιλείας. Έχουμε κάνει κάποια βήματα και σε επίπεδο τραπεζικής ένωσης, αλλά τα συμπεράσματα δεν τα έχουμε βγάλει ακόμα. Και υπάρχει ένα θέμα το οποίο με ανησυχεί. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα έλεγα γεννιέται σε επίπεδο λογιστικών κανόνων. Η άνοδος του βάρους των συντονισμών, των δομών, των διεθνών οργανώσεων. Μιλάμε για ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι ουσιαστικά καθορίζουν την δημόσια ημερήσια διάταξη. Αυτό το θέμα της, ε, της λήψης αποφάσεων για το ενιαίο ε, των λογιστικών κανόνων είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει και μία κάποια θα έλεγα ε, στενή σχέση ανάμεσα στο EISB και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ίσως ή κάποιο άλλο διεθνές αναγνωρισμένο όργανο. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε από τον οργανισμό αυτό το Monitoring Group, κάτι το οποίο στην ουσία κόβει την ανάγκη, διακόπτει την έκφραση της ανάγκης επικοινωνίας με έναν ε, ευρύτερο και αναγνωρισμένο διεθνή δημόσιο οργανισμό. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα παρακολουθήσουμε στενά. Δεν ξέρω, αυτές οι οργανώσεις είναι νέες οργανώσεις, είναι οργανώσεις που πρέπει να έχουν σχέση με το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, δεν ξέρω να πω εδώ τίποτα. Αλλά το θέμα της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα το οποίο θέτει και τη συμμετοχή μας στην διάρθρωση των οργανισμών αυτών των διεθνών. Έχω μια επιπλέον ανησυχία ε, βλέπουμε ότι οι διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες οργανώνονται επί τη βάση των δικών τους συμφερόντων, αγνοώντας ε, τα παγκόσμια διακυβεύματα σε επίπεδο χρηματοπιστωτικής ισορροπίας ή σε επίπεδο κατανομής πόρων ακόμα περισσότερο. Μάλετιτς Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Σιλβή για την πρωτοβουλία της. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον των διεθνών χρηματοπιστωτικών φορέων. Η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν ασκήσει πίεση για διαθετικές μεταρρυθμίσεις, έχουν χρηματοδοτήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και έχουν δώσει δανειοδοτήσεις ιδιαίτερα ευνοϊκές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίζει τη δράση της με τους φορείς αυτούς, να λαμβάνει υπόψη μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο την ε, σύνδεση με τους φορείς αυτούς και αυτά να αντανακλώνται και στην ε, στάση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα κρατημέλη. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και αυτό είναι πολύ θετική αυτή η έκθεση και χαιρετίζω την ύπαρξή της. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η συγγετρία για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Πάρα πολύ σύντομα Ακόμα και αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, σας ευχαριστώ όλους για το επικοδομητικό σας πνεύμα από όλες τις πλευρές. Δεν είχαμε τον εισηγητή της ΓΚΟΕ, αλλά φυσικά θα το συναντήσω και στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θέλησε να επιληφθεί αυτού του θέματος που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλέ παρατηρήσει οι οποίε είναι πολύ ενδιαφέρουσε για μένα, αλλά βλέπω να υπάρχουν σημεία σύγκληση μεταξύ του. Είναι πολύ σωστό το είπε η κυρία Πιετικάινεν, η κυρία Νεύρογκ, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε προδραστικοί. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δημοκρατία δεν είναι μονάχα ο έλεγχος εκ των υστέρων, αλλά είναι ενδεχομένως και η ικανότητα να δίδουμε ενάρχηματα και κατευθύνσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να κάνουμε και τα δύο. Δεν πρόκειται λοιπόν τόσο πολύ για το να προασπίσουμε το κύρος και την επιρροή του Κοινοβουλίου, όσο το να προασπίσουμε τις αξίες μας. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε λανθασμένους αγώνες. Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε περισσότερες εξουσίες, απλώς προσπαθούμε να είμαστε υπόλογοι σε αυτούς οι οποίοι μας έφεραν εδώ. Και εγώ συμφωνώ με τον Σφεν Γκίγκολ, ότι πρέπει να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Φόξ δύο φορές χρησιμοποίησε το βρετανικό χιούμορ, του οποίου είναι εξαίρετος ε, εκπρόσωπος. Ιδίω όταν αναφέρθηκε στον πραγματισμό μου. Ελπίζω όμω ότι και οι Βρετανοί θα δείξουν τον ίδιο πραγματισμό στη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση η οποία δεν πρέπει να είναι ιδεολογική. Τούτου λεχθέντο δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ε, αφελεί. Έχουμε πράγματι κάποια συμφέροντα τα οποία πρέπει να υπερασπιστούμε. Δεν είναι λάθο οι Ευρωπαίοι να το πράττουν αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιώντα την ισχύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την κοινή δράση. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε το ίδιο νόμισμα, κάτι το οποίο δεν θέλησαν οι Βρετανοί να κάνουν, δείχνει, μάλλον οδηγεί τις άλλες χώρες σε κοινά συμφέροντα και την ανάγκη να σεβαστούν μεν τους εταίρους τους που δεν είναι στη ζώνη ευρώ, αλλά συγχρόνως να μην υποτιμήσουν την ανάγκη κοινής δράση στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό και την υπεράσπιση του ευρώ. Αυτό είναι προς το γενικό συμφέρον, δεν είναι μονάχα προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και προς το παγκόσμιο συμφέρον να έχουμε ένα νόμισμα το οποίο συμβάλλει στην παγκόσμια σταθερότητα και όπως ελέγχθη πολύ σωστά μπορεί να εξασφαλίσει μέσα στην ε, πολυμορφία των κρατών μελών σε κοινέ θέσει. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να καταδείξουμε και πάλι ότι μία από τι βασικέ αρχέ των συνδικών που πολλέ φορέ χάνεται από τα μάτια μα είναι ότι πρέπει να υπάρξει ο λεγόμενο έντιμο η λεγόμενη έντιμη συνεργασία μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργασία προς το κοινό συμφέρον. Να μην δρούμε δηλαδή με τρόπο που αντιβαίνει προς τα συμφέροντα των άλλων χωρών. Αυτό το οποίο με ενοχλεί μερικέ φορέ δεν είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τα εθνικά κράτη, αλλά ότι ορισμένε φορέ βλέπουμε σε κάποιου φορεί να υπάρχει το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο. Δηλαδή γίνεται μια διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα κείμενο. Κάποια χώρα βρίσκεται σε μειοψηφία στι διαπραγματεύσει και καταφεύγει στα διεθνή φόρα για να μπορέσει να ανατρέψει αυτό που αποφασίστηκε στα ευρωπαϊκά όργανα. Υπάρχουν κάποια κράτη, εγώ ξέρω κάποιο συγκεκριμένο κράτος που ορισμένες φορές κάνει τέτοιες ενέργειες. Δεν λοιπόν πρέπει μονάχα να κατηγορούμε τους άλλους, αλλά να καταλάβουμε ότι έχουμε κοινέ δεσμεύσεις, κοινέ υποχρεώσεις και δεν μπορούμε να τα συνοψίσουμε όλα αυτά με το να είμαστε μαζί όταν μας βολεύει και όταν δεν μας βολεύει να έχουμε τελείως αποκλήσεις και διαφορετικές απόψεις έναντι των ε, έξω χωρών. Αυτό ελέγχθη για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένα θέμα. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα εκεί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται με διαφορετικό τρόπο. Έχουν λάβει πολλές ε, εξελίξεις χώρα τα τελευταία χρόνια που ίσως δεν τις βλέπουμε γιατί είμαστε εστιασμένοι στο καθημερινό επίπεδο αλλά υπάρχει μια, υπάρχει μια διεθνοποίηση για όλα αυτά τα θέματα και εξετίμησε ιδιαίτερα αυτό που είπε και ο Σβέν Γκίνγκολτ. Πρέπει να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτά τα οποία κάναμε στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι περιορισμένα, αλλά είναι ο μόνος χώρος στον κόσμο όπου μπορούμε να έχουμε και συνεργασία και δημοκρατία. Όχι μονάχα δημοκρατία, αλλά και κράτο δικαίου, γιατί δεν έχουμε μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η ύπαρξη δημοκρατικών φορέων που προσδίδουν την ε, ε, νομιμοποίηση, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει και η δυνατότητα νομικής προσφυγής. Η Ευρώπη λοιπόν έχει δείξει ένα παράδειγμα στον τομέα αυτό. Αυτοί με τους οποίους έχω μιλήσει σε αυτούς τους διεθνείς φορείς επιβεβαιώνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ο δρόμος της Ευρώπης είναι ένα παράδειγμα για να μπορέσει να εξασφαλιστεί περισσότερο κράτο δικαίου εκεί που προς το παρόν υπάρχουν μονάχα ισορροπίες ισχύω. επομένω πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε τη Σιλβί Γκουλάρ που μας υπενθύμησε και την αρχή της συνεργασίας που κατοχυρώνονται στις ε, συνθήκες. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει εξέταση. Ναι, συγγνώμη πρόεδρε που σας διακόπτω, αλλά άκουσα αυτά που είπαν κάποιοι από τους κοιόδης. Αν χρειαζόμαστε πιο πολύ χρόνο, καταρχάς επειδή είχαμε αυτά τα σημαντικά έγγραφα, τις μελέτες, ακόμα και το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό που λέτε, ήθελα να σας πω ότι ως εισηγήτρια είμαι πρόθυμη να δώσω πιο πολύ χρόνο εφόσον αυτό χρειάζεται, αλλά φυσικά αυτό το αποφασίζει και ο Πρόεδρος και οι συντονιστές. Ο Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα για να προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα. Αν υπάρχει τέτοιο αίτημα από την εισηγητρία και τους κοιόδης. 15-16 Ιουλίου τώρα προβλέπεται η εξέταση του κειμένου και για το Σεπτέμβριο για τις ε, τροπολογίες προθεσμία. Αν μετά από τις μελέτες αυτές θεωρείτε ότι χρειάζεται πιο πολλής χρόνος, θα σας ενημερώσουμε για τις ενδεχόμενες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Ευχαριστώ και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Εξέταση των τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Μπάγε για την ε, έκθεση της ΔΕΒΕ για τη φόρο διαφυγή και φόρο αποφυγή ως προκλήσεις για την διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα θέμα κρίσιμο και συμπληρωματικό ασφαλώς προς το έργο που κάνουμε εδώ και στην Επιτροπή Τάξη. 98 τροπολογίες λάβαμε και δίνει το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ηγητές για την ποιότητα τη συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει κατά τη διάρκεια της εργασία αυτή τη έκθεσης. Ο στόχος ήταν να φτάσουμε στην ευρύτερη δυνατή συνένεση. Βέβαια, έρχεται σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως το LuxLeaks και άλλε περιπτώσεις φοροαποφυγής που έχουν γίνει γνωστές. Πρέπει όμω να δώσουμε προτεραιότητα στην ε, φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε πώ δρούμε κατά τη φοροαποφυγή και να βοηθήσουμε και τι αναπτυσσόμενε χώρε και αυτέ με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουν την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Χρήματα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την υγειονομική περίθαλψη, την παιδεία, τι κοινωνικέ παροχέ, πολλέ φορέ χάνονται λόγω τη φοροδιαφυγή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καθορίσουμε σαφώ τι είναι ο φορολογικός παράδεισος, να υπάρχει μια σαφής δυνατότητα ορισμού ώστε να καταρτήσουμε και κάποιο κατάλογο των φορολογικών παραδείσων, μια μαύρη λίστα για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε κατά του φαινομένου πρέπει να μιλάμε όλοι με την ίδια γλώσσα. Επίση πρέπει να έχουμε και μια κοινή φορολογική βάση φορολογία των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο να είναι <clears throat> υποχρεωτικό καταρχήν για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε και τι συνεργατικέ ευρωπαϊκέ εταιρείε και να προχωρήσουμε σε φορολογική εναρμόνιση στο βαθμό του τεχνικά αφικτού για τις επιχειρήσεις. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευκυβερνησία και την συνεργασία για τα φορολογικά θέματα με τρίτες χώρες και έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να εφαρμόζονται οι κανόνες της <clears throat> αποφυγής διπλής φορολογίας. Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν αυτούς τους κανόνες για να μειώσουν τη φορολογία τους ακόμα και προς το μηδέν, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και επίσης ζητούμε από την Κομισιόν <clears throat> να δημιουργήσει μια οδηγία κατά της αποσύνδεσης μεταξύ του χώρου δραστηριότητας μιας εταιρείας και του χώρου όπου φορολογούνται τα κέρδη για το στόχο της φοροαπαφυγής. Θέλουμε επίσης να δημιουργηθεί ένας ε, ένα παγκόσμιο σύστημα για να συνδέει όλες τις χώρες για την ε, παροχή αναφορών για τη φορολογική κάλυψη και να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν να υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν σε μια πιο δίκαια εξισορρόπηση της φορολογίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα για το ΕΛΚ. Ο Τόμ Φαντεκαριλάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία Νομίζω ότι ο συμβιβασμό ε, που εξετάζεται είναι καλό μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών θέσεων για τα ειδικά θέματα σε ό,τι αφορά τι συστάσει ανά χώρα. Βρήκαμε ένα καλό συμβιβασμό με την εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την περιορισμό των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων. Κάποια πράγματα δεν μας βρίσκουν σύμφωνος και θα ζητήσουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Καταρχάς, το θέμα για την ελάχιστη τιμολόγηση, για ελάχιστο συντελεστή για ε, εταιρική φορολόγηση. Εδώ είναι το θέμα αυτό διαπραγμάτευτο για μας. Επίσης, θέλουμε να υποστηρίξουμε τον ορισμό ε, των προλογικών παραδείσων για να προωθήσουμε και το έργο του ΑΣΑ που έχει κάνει προς την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύω ειλικρινά ότι πρόκειται για μια ισορροπημένη γνωμοδότηση και πραγματικά ευχαριστώ τον εισηγητή για τον εκτό πνεύμα που έδειξε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Η Μπέτεξ Ja, ähm, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία κύριε Μπαγιέ. Για το ECR να τονίσω τα θέματα αυτά που δεν μας βρίσκουν ε, σύμφωνους, όπου έχουμε διαφορετική άποψη. Το γενικό πνεύμα είναι ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές ε, και η φορολόγηση γενικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες δηλαδή θα πρέπει να εξισωθούν με τις αναπτυγμένες χώρες σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος ως σειρά. Πιστεύω ότι οι αναπτυσσόμενες χώρα καταρχάς θα πρέπει να, να δημιουργήσουν κάποια ε, δικαιώματα ε, ιδιοκτησίας, να φροντίσουν να μην υπάρχει διαφθορά, ε, χρηματοοικονομικές ιδρύματα ανεξάρτητα δικαστηρία. Όταν θα έχουν εισηχθεί και εφαρμοστεί όλα αυτά τα στοιχεία, τότε στη συνέχεια έχει νόημα να αυξηθεί κάπως ο φορολογικός συντελεστής για να υπάρχει μια βασική α, χρηματοδότηση όλων αυτών των στοιχείων που δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση στις αναπτυσσόμενες χώρες και για να ενισχυθούν και οι επενδύσεις από την αλλοταπή και οι εγχώριες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος πρώτα να, αυξηθούν η φορολογία, να αυξηθεί η φορολογία, να γεμίσουν τα ταμεία και μετά να γίνουν αυτές οι αισθαντικές αλλαγές. Είναι λάθος η σειρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα για την άλλη, ο κύριος Γεζίκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και εγώ για τη δουλειά του. Ήταν φιλόδοξη η προσέγγιση του. Προσπάθησε σκληρά να πετύχει την πιο ευρεία δυνατή συνένεση. Είναι αρκετά ξεκάθαρη η γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι περιέχει ένα καλό βαθμό φιλοδοξίας, λαμβάνει υπόψη της ε, ιδιαιτερότητας των αναπτυσσόμενων χώρων και αυτό αποτελεί κάτι που είναι βασικό για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στις χώρες αυτές. Τα βασικά στοιχεία της έκθεσης ε, λίγο πολύ παρουσιάστηκαν ήδη. Εγώ απλά να πω ότι χαίρομαι που καλεί στο κείμενο ο εισηγητής να υπάρχουν ίσοι όροι ανταλλαγή πληροφοριών και πιλωτικά project, πιλωτικά έργα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν στον τομέα αυτό, καθώς, τα καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν απαραίτητα πάντα πόρους προς την κατεύθυνση αυτή. Το κείμενο επίσης ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει την αρχή ότι οι πολυεθνικές εταιρείε θα πρέπει να κάνουν εκθέσεις αναχώρα για όλους τους κλάδους ενώ παράλληλα διασφαλίσει δεν θα αυξηθεί το γραφειοκρατικό άκθος για τις μικρομεσαίες. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι αρκετά ισόρροπη, φιλόδοξη η έκθεση συνολικά και νομίζω ότι με άμεση μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Νικού, ε, τη βλέπω πουθενά. Η Εύα Ζολή για τους πράσινου. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα της παρουσίασής του και για την ευαισθησία την οποία έχει επιδείξει. Είναι από τα πρόσωπα τα λίγα που έχουν καταλάβει ότι η φορολογία των πολιεθνικών συνδέεται με την ανάπτυξη των χωρών σε περιοχές όπως της Αφρικής. Εμείς είχαμε κάνει μία συνάντηση με τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες και διαπιστώσαμε πόσο δεν γνωρίζουν ε, το τι συμβαίνει στον κόσμο και πόσο προασπίζονται το θέμα της φορολογίας, της βέλτιστης μορφής φορολόγησης για τις επιχειρήσεις τους με τελικό στόχο το να μην πληρώνουν καθόλου φόρο και τι συνέπειες έχει αυτό στον κόσμο. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για αυτήν την γνωμοδότηση η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους. και όπως λέτε και εσείς στις συμβιβαστικές προτάσεις σας εμείς προτείνουμε μια ενιαία μορφή φορολογίας ε, των επιχειρήσεων και ένα ελάχιστο ποσοστό φορολογίας επίσης. Έχει εκφραστεί η επιθυμία του Κοινοβουλίου επανειλημμένα να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον δικό της κατάλογο σε εισαγωγικά των λεγόμενων φορολογικών παραδείσων υποστηρίζετε εσείς την καταγραφή της κατάστασης σαν αναπολιεθνική και θα συμφωνήσω μαζί σας αύριο στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γύρω από το θέμα των δικαιωμάτων των μετόχων. Ε, το θέμα αυτό θα συμπεριληφθεί στη συζήτηση. Επίσης νομίζω ότι θα γίνει δεκτή και η τροπολογία σας υπαρήθμε 63, διότι ζητά να υπάρξει ε, μία σε βάθος αλλαγή και μεταρρύθμιση του εταιρικού δικαίου και να καταργηθεί η δυνατότητα χρήσης τεχνητών εταιρικών δομών με μοναδικό στόχο τη φορολογική διευκόλυνση, κάτι το οποίο έχει τρομακτικές συνέπειες στις υποανάπτυξη χώρες. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής έχει πάλι το λόγο. Α, συγγνώμη, ο κύριος Μαριάς έχει δει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλά κράτη διότι δεν μπορούν να αποκτήσουν έτσι δημόσια έσοδα. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν βεβαίως να επενδύσουν τα ποσά αυτά στις δημόσιες δαπάνες, κυρίως στην ε, παιδεία, στην ε, υγεία. Αυτό ισχύει για πάρα πολλές χώρες, ισχύει και για την Ελλάδα. Υπάρχουν ε, τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες ολιγάρχες με διάφορες offshore εταιρείε και φορολογικούς παραδείσους με στόχο πραγματικά την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Και αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην πατρίδα μου την Ελλάδα, διότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εσόδων. Το δεύτερο θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε ένα φορολογικό ανταγωνισμό, καθώς δίνουν με τον β τρόπο ευκαιρίες σε κάποιες πολυεθνικές κυρίως να εγκατασταθούν σε αυτά τα κράτη και έτσι να φόρο αποφύγουν να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους σε άλλες χώρες. Είχαμε την περίπτωση των LuxLeaks την οποία διερευνούμε. Το τρίτο θέμα που πρέπει να δούμε είναι οι ενδοομιλικές συναλλαγές. Διότι εάν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, πραγματικά θα υπάρχει μια συνεχής φοροδιαφυγή και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ενδεχόμενα ένα συνεχής φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Επομένως πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις όπου τα κέρδη των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων να φορολογούνται εκεί όπου πραγματικά δημιουργούνται. Εκεί όπου οι πολυεθνικές πραγματικά δημιουργούν τα κέρδη. Να μην έχουμε δηλαδή αυτή την τεχνική των ενδοομιλικών συναλλαγών και να έχουμε αυτή την φοροαποφυγή. Νομίζω ότι αυτά είναι τρία βασικά συστήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει με κάποιο τρόπο η εισήγηση η οποία παρουσιάστηκε και είναι θέματα τα οποία πρέπει πραγματικά να τα αντιμετωπίσουμε σε βάθος. Διαφορετικά θα έχουμε μία διαδικασία με φορολογικούς παραδείσους, με περιοχές όπου θα γίνεται συνεχής φοροδιαφυγή, και αυτό βεβαίω είναι ει βάρο της ίδιας της ανάπτυξης των χωρών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μαριά, θα συμφωνήσω σε πολλά πράγματα αλλά το θέμα είναι ποια είναι η γνωμοδότηση, η άποψη μάλλον της Επιτροπής μας απέναντι στην προβληματική των χωρών των υποανάπτυξη. Και γι' αυτό συνεχίζουμε τη μέθοδο αυτή reporting αναχώρα έτσι ώστε να πείσουμε ότι η φορολογία θα πρέπει να πληρώνεται εκεί όπου επιτελείται η δραστηριότητα και η εργασία περιμένουμε και τι μέτρα θα προτείνει η συγκεκριμένη επιτροπή για τα φορολογικά με τις ειδικέ φορολογικές ε, ρυθμίσεις. Χρειάστηκε να κάνουμε μια συμβιβαστική πρόταση, πάντως αυτό πρέπει να καταλάβετε. Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε τις απόψεις όλων των συναδέλφων, ελπίζω να υπεψηφιστεί το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε πράγματι το απόγευμα την έκθεσή σας και ε, στην αρμόδια επιτροπή της στην 1η Ιουνίου. Επόμενο θέμα. Στατιστική για το ισοζύγιο πληρωμών, διεθνείς εμπορικές υπηρεσίες και άμεσες ξένες επενδύσεις. Εξέταση της έκθεσης. Ο Σβεν Γκίγκολντ είναι ο εισηγητής, έχει το λόγο. Chair, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συνοδεύτους για την παρουσία τους και τη συμβολή τους σε αυτήν την τόσο συναρπαστική έκθεση. Ο κανονισμός που αφορά την, το ισοζύγιο πληρωμών της Διεθνής Χρηματοπιστωτικής Υπηρεσίας και στατιστικές είναι τμήμα του Γενικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Η παραγωγή στατιστικών που να έχουν αξιόπιστο χαρακτήρα στους τομείς αυτούς για την παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών ροών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα των οικονομικών πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι κατευθυντικέ γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με τι νομικέ υποχρεώσει που απορρέουν από το πλαίσιο ευκυβερνησία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα οικονομικά θέματα. Οι στατιστικέ αυτέ λοιπόν είναι απαραίτητε για την παρακολούθηση και την εποπτεία που θεσπίζεται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μετά από την έγκριση του αρχικού κανονισμού και την εφαρμογή του, οι διεθνεί χρηματοπιστωτικές βάσεις έχουν εντατικοποιηθεί και αυξηθεί η πολυπλοκότητά του. Η χρησιμοποίηση ειδικών χρηματοπιστωτικών φορέων για την ε, διοχέτευση χρηματοπιστωτικών ροών έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την παρακολούθηση αυτών των ροών και δεν εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ανιχνευσιμότητα και τον κίνδυνο πολλαπλής λογιστικής καταπικόνησης. Ο αγώνας κατά της ε, φοροαποφυγής λοιπόν και τη επιθετική πολιτική σχεδιασμού στα φορολογικά παραμένει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό ο κανονισμός 184 του 2005 θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να αντιμετωπίσουμε ένα διπλό στόχο. Πρώτα απ' όλα, η νομοθετική πρόταση τη Κομισιόν είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να αυξήσουμε τη διαφάνεια και την ε, λεπτομέρεια των στατιστικών που έχουν να κάνουν με το παγκόσμιο εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές ροές και επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πρόσφατες νομικές ε, ρυθμίσεις για να είναι πιο χρήσιμα αυτά τα στοιχεία για πολιτικές αποφάσεις. Και όπως είπε και η Κομισιόν στην νομοθετική της πρόταση, ο κανονισμός θα πρέπει να επικαιροποιηθεί για να εξασφαλίσουμε ότι συνάδει με τους κανόνες του, ε, της Συνδίκης Λισαβόνα σε ό,τι αφορά τις κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις που είναι στη διάθεση της Κομισιόν. Εγώ πιστεύω ότι η διαφάνεια και η λεπτομεριακότητα των ε, διαδικασιών αυτών μπορεί να αυξηθεί με την αύξηση των ε, υποχρέωσεων παροχής εκθέσεων ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των χρηματοπιστωτικών ροών όπως αναφέρεται στο τροπολογίες 19, 20 αλλά και 21 που δίδουν ορισμένες τεχνικές προσαρμογές για το παράδειγμα 1 χωρίς, χωρίς να δημιουργούν πρόσθετο άχθος σε στατιστικό επίπεδο. Όπως προτείνεται λοιπόν από την τροπολογία με 12, ο γενικός στόχος της αύξησης της ε, διαφάνειας και ανιχνευσιμότητας μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα αν το νέο νομοθετικό πλαίσιο λάβει υπόψη τρεις πρόσφατες χειροτομίες Πρώτα απ' όλα, ο εντοπιστής για τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό φορέα που χρησιμοποιείται για να ε, εντοπίζονται καλύτερα οι χρηματοπιστωτικές ροές. Η αρχή του τελικού δικαιούχου που εμφανίζεται στην οδηγία κατά της έκπλησης χρημάτων και τρίτον η βάση δεδομένων που βρίσκεται στην συντονισμένη ε, πρωτοβουλία για τις επενδύσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε καλύτερα στατιστικά στοιχεία, έχω προσθέσει και ορισμένε τροπολογίες. Η τροπολογία 14 προβλέπει ότι στατιστικές οι οποίες συντάσσονται ε, μέσα στον κανονισμό αυτό θα πρέπει να κάνει μια διάκριση μεταξύ άμεσης ξένης επένδυσης και επενδύσεως που προέρχεται από συγχώνευση επιχειρήσεων και αυτών οι οποίες δεν αυξάνουν το κεφάλαιο κίνησης του φορέα ο οποίος υπέστη αλλαγή ιδιοκτησίας. Τροπολογία 13. Ενισχύει την συνεργασία της Κομισιόν με τη Eurostat και άλλους φορείς διεθνούς, διεθνού, διεθνούς χαρακτήρα ώστε να καλύπτονται όλες οι στατιστικές πηγές που αφορούν και αυτόν τον κανονισμό, όπω είναι ο ΣΑ και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να προωθηθεί η καλύτερη μεταλαμβάνευση εμπειρογνωμοσύνη και θα αυξηθεί και η ποιότητα των στατιστικών σε σχέση με το ισοζυγείο πληρωμών. Η τροπολογία 18 προβλέπει ότι η Eurostat θα πρέπει από μία πλευρά να βελτιώσει την ποιότητα των στοιχείων που αφορούν το, ε, το ισοζύγιο πληρωμών και των επενδύσεων και επίσης, όπως είπατε στις φαρχικές μου παρατηρήσεις, θα πρέπει να υπάρξει επιγράμμιση αυτού του κανονισμού με τα, τις πρόνοιες της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό λέει και η τροπολογία 10. Η συνθήκη της Λισαβόνας πράγματι κάνει μία διάκριση μεταξύ κατεξουσιοδότηση πράξεων που η Κομισιόν μπορεί να χρησιμοποιήσει για να τροποποιήσει μερικά δευτερεύοντα δευτερεύουσα σημασία στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 291, και συγχρόνως των εφαρμοστικών εξουσιών η Κομισιόν, όταν πρόκειται για να θεσπιστούν νομιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή δεσμευτικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέει το άρθρο 92. Οι προσδιορισμοί των χρηματοπιστωτικών ροών δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι δευτερεύοντα στοιχεία τα οποία μπορούν να τύχουν τροποποίηση από την Κομισιόν. Είναι στοιχεία όμως τα οποία έχουν να κάνουν με την καρδιά τη ρύθμιση. και τα στοιχεία αυτά λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρούνται με την νομοθετική διαδικασία η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τους δύο συνομοθέτες. Με τον ίδιο τρόπο μία έκθεση για την ποιότητα της ε, νομοθεσίας δεν είναι ουσιώδες στοιχείο. Στην διαδικασία τροπολογιών και τροποποίησης θα πρέπει να ξεπεράσουμε το, την εμβέλεια της έκθεσής μου και να λάβουμε υπόψη τις εκθέσεις ποιότητας και τα πρότυπα ποιότητας τα οποία τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο του ουσιώδης. Όλα αυτά αναφέρονται τις τροπολογίες για τις ε, αιτιολογικές σκέψεις. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα καταλήξει μια γενική προσέγγιση. Σύντομα όμως θα το πράξει και η έκθεσή μου ευθυγραμμίζεται με το Συμβούλιο στις εξή πτυχές. Η υποχρέωση για την Κομισιόν να ζητά την άποψη της CMFP, της Επιτροπής για τις Στατιστικές Χρηματοπιστωτικού Χαρακτήρα και Ισοζυγίου Πληρωμών για όλες τις υποθέσεις που είναι στην αρμοδιότητά. Δεύτερον, το να μειωθεί η εμβέλεια των πράξεων κατά εξοδότηση της Κομισιόν, ώστε να μην αλλάζουν το βασικό ενοιολογικό και στατιστικό πλαίσιο. Και τρίτον, η κύρια διαφορά μεταξύ της έκθεσής μου και της άποψης του Συμβουλίου είναι ότι το Συμβούλιο δεν θέλουν να τροποποιήσουν το παράδειγμα 1. Θέλω να κλείσω με μια γενική παρατήρηση. Αυτή η στατιστική έκθεση και εδώ συνεργαστήκαμε με τους σκιώδεις εισηγητές και βρήκαμε πολύ ενδιαφέρουσες συγκρούσεις μεταξύ των εθνικών στατιστικών φορέων, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τις Εθνικές Τράπεζες, Κεντρικές Τράπεζες και την Κομισιόν. Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε μια συνεδρία στην παρουσία των σκιωδών και του προσωπικού τους μεταξύ των αντιμαχωμένων πλευρών για να βρούμε μια λύση. Δεν καρποεφόρησε αυτή η προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο τώρα θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια θέση για το θέμα αυτό και ελπίζω για την υποστήριξη όλων των σχιωδών και πιστεύω ότι στο τέλος θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία θα εξασφαλίσει στατιστικές ποιότητος για όλους αλλά συγχρόνως θα εδραιώσει και τις δημοκρατικές αρχές. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι μια σαφή, σαφής ευκαιρία για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να ακούσω και τις απόψεις των σκιωδών και τονίζω ότι δεν είναι μια έκθεση η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε πολιτικές αντιπαραθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και για τα καταληκτικά του σχόλια. Ξέρουμε ότι είναι περίπλοκη η δομή της συνθήκης για τα διάφορα δικαιώματα στο στατιστικό κλάδο και ότι όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες στην κατάσταση της σχετικής νομοθεσίας. Προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία. Για να βρούμε μια καλή λύση όπως κάναμε και στο Γενικό Κανονισμό για τα θετικά στοιχεία. Δεν έχει έρθει ο σκιώδης ε, του EPP, του ΕΛΚ, οπότε δεν είναι το λόγο σε πάνω από Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σβέν και Γκόλτ. Εξετίμησα διόντως την ισορροπία που χαρακτηρίζει την πρόστασή του και θα ήθελα να πω ότι μετά την ομιλία μου ζητώ συγγνώμη, πρέπει να φύγω γιατί είμαι εισηγήτρια στην άλλη μου επιτροπή και δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη συζήτηση μέχρι τέλους. Κάποια μικρά σχόλια σε σχέση με αυτά τα οποία μας είπε ο Γκίγκολτ, σύντομα. Κάποιες γενικές σκέψεις πρώτα. Το θέμα αυτό δεν θα προκαλέσει τεράστιες πολιτικές συζητήσεις στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων. Είναι όμως αλήθεια ότι το να έχει κανείς αξιόπιστες στατιστικές είναι ένα χρήσιμο μέσο για να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα των οικονομικών πολιτικών και του σεβασμού, της επαλήθευσης του σεβασμού των υποχρεώσεων που προέρχονται από την κοινή διακυβέρνηση στα πλαίσια της καταπολέμησης των μακροπρόθεσμων ανισοτήτων όπως επίσης και η πλήρης διαφάνεια στις στατιστικές αυτές πηγές είναι χρήσιμο για την καταπολέμηση της ανακύκλωσης του ε, χρήματος όπως επίσης και των φορολογικών απατών. Ε, επί της ουσίας τώρα, <clears throat> στα θέματα τα οποία ε, τίθενται στην έκθεση, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο αυτά τα οποία θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά και στα οποία συμφωνώ με τον Γκίγκολτ ανάγκη ε, ε, σαν παράδειγμα ε, της, του καθορισμού της υποχρέωσης δημοσίευσης στοιχείων, της χρήσης νέων καινοτόμων μεθόδων στα πλαίσια της ροής των κεφαλαίων, διεθνής καταγραφή της νομικής προσωπικότητας των οικονομικών οντοτήτων, όπως επίσης και δεδομένα των τραπεζών για τις άμενες επενδύσεις. Είναι επίσης χρήσιμο να υπογραμμίσουμε εδώ την ανάγκη που υπάρχει για μια ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Εροστάτα και τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς. Ήμουν παρούσα στην επικοδομητική συνάντηση η οποία οργανώθηκε ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση και την Επιτροπή. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε στο τέλος της παρουσίασής του ο κύριος Γκίγκολτ Απ' τη μία θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στις ανησυχίες που υπάρχουν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών. Και από την άλλη θα πρέπει εμείς να διατηρήσουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε μια πραγματιστική απόπειρα έβρεση των κατάλληλων λύσεων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μέσων τελικά, μέσα τα οποία θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους κεντρικούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο ή μάλλον δεν βλέπω κάποιους άλλους σκιώδες. Από, την, από τους φιλελευθέρους θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο εξ του κ. Τόρβαλτς. Όχι. Λοιπόν, είναι... Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Eurostat και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Ντάβιλα για την Eurostat. Όχι. είμαι υπεύθυνη στα θέματα των στατιστικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντική η έκθεση του κ. Γκέγκολτ. Υπογραμμίζει σωστά τη σημασία που έχει ο κανονισμός εμείς προτείνουμε να τροπολογήσουμε τον κανονισμό για τις υπηρεσίες αυτές και για τις στατιστικές σχετικά με τις άμεσες επενδύσεις. Στόχος είναι η εναρμόνιση του κανονισμού αυτού με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε μετά από τις συνθήκες Λισαβόνας θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει την δυνατότητα έκδοσης εξουσιοδότηση πράξεων και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να λάβει υπόψη και τις νέες ρυθμίσεις για τα ποιοτικά επίπεδα τα οποία απαιτούνται στα πλαίσια αυτών των στοιχείων. Είμαστε στη διάθεσή σας πάντως στο μέλλον για περαιτέρω συνεργασία και για περισσότερες διευκρινήσεις. Δεύτερος στόχος της πρότασης, την οποία κάναμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να ευθυγραμμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις της Επιτροπολογίας εφαρμόζονται με τον πρόσφατα αναθεωρισμένο κανονισμό 223. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι είναι θετικές οι προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση Giggold. Έχουμε κάνει μια πρώτη αξιολόγηση των τροπολογιών σχετικά με τις ε, ε, τροπολογίες για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και έχουμε ήδη σημειώσει ότι η επιθυμία που εκφράζεται για την αύξηση των δεδομένων στοιχείων είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει θετικά την ποιότητα των στατιστικών. Θα συνεχίσουμε όπως είπα να συνεργαζόμαστε γιατί κάποιες από αυτές τις προτάσεις ε, διευκρινίζουν καλύτερα τον κανονισμό αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε επίσης και επικαλύψεις, γιατί κάποια από τα δεδομένα αυτά έτσι και αλλιώς είναι διαθέσιμα. Συμπερασματικά λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Γκίγκολτ, γιατί εξέτασε σε βάθος το θέμα του και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί του. Σας ευχαριστώ και τώρα να στραφούμε προς τον κύριο Μπύρα από την ΕΚΤ. Ευχαριστώ πολύ υποστηρίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική θέληση πίσω από την πρόταση και το σχέδιο του κειμένου του εισηγητή. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τρία τμήματα, τρεις ενότητες. Καταρχάς, οι πολλέ ενδιαφέρουσες ιδέες για τις άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις, ό,τι αφορά και την συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συστήματος Στατιστικών Στοιχείων και Κεντρικών Τραπεζών για το πρώτο θέμα, γιατί σε πέσει άμεσες επενδύσεις. Έχουμε τρεις προτάσεις που ήδη έχει παρουσιάσει ο εισηγητής ε, για τις αντικεφαλαιοκές ε, ροές ε, βάσει των κριτηρίων δικαιούχου αυτό μπορεί να αυξήσει την αναλυτική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σωστικών στοιχείων και μπορεί να συμβάλλει και στην διαφάνεια και την ανεχνευσιμότητα των χρηματοοικονομικών ροών, όπως, εξετε, εξηγείται στο επεξηγηματικό σημείο μας. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι πληροφορίες, η συλλογή των πληροφοριών είναι πολύ πιο περίπλοκη λόγω των αλλαγών και λόγω των διαφορετικών διεθνών ε, δικαιοδοσιών για να υπάρξει δηλαδή συλλογή όλων αυτών των συζητικών στοιχείων πρέπει να υπάρχει συνεργασία με άλλα διεθνή σώματα, ο g Για το λόγο αυτό μπορεί η ροή αυτή πληροφοριών να πρέπει να αναφέρεται μετά μια απομεταβατική περίοδο μεταξύ των διαφόρων ε, διεθνών φορέων Δεύτερο στοιχείο για τις αλλοδαπές άμεσες επενδύσεις. Τα στατιστικά στοιχεία θα δώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και ανιχνευσιμότητα των αλλοδαπών επενδύσεων και δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένο κόστος για τα κρατημέλη. που πολλές εξ αυτών υποστηρίζουν έτσι και αλλιώς τις προτάσεις ε, για του Διεθνέ Νομισματικού Ταμείου. Τελευταία πρόταση στο πλαίσιο αυτό. Διάκριση μεταξύ takeover και greenfield επενδύσεων. Πολύ χρήσιμο τομέα για να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο των άμεσων αλλαταπών επενδύσεων. and more conceptual work. Και χρειάζεται όμως και πολλή δουλειά προτού επιλέξουμε αυτή την προσέγγιση για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα είναι επαρκώς συγκρίσιμα. Άρα, συνολικά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή. Υποστηρίζουμε, την υποστηρίζουμε πολιτικής άποψης, απλά παρατηρούμε ότι η εφικτότητα και η εφαρμογή θα προαπαιτούσε στενή διεθνή συνεργασία και ενδεχομένω δεν μπορεί μόνο της Ευρωπαϊκή Ένωση να τα περάσει αυτά. Άλλες δύο παρατηρήσεις για τη διαδικασία σε ό,τι αφορά την ε, νομοθετική αυτή πρόταση. Σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές αρμοδιότητες, εδώ πέρα εκτιμούμε αυτά που αναφέρει στο επεξηγηματικό σημείωμα ο εισηγητής, ότι οι αναθεωρήσεις ε, των στοιχείων αυτών όπου περιλαμβάνονται στο παράδειγμα 1 δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μη ουσιώδες στοιχείο αλλά στοιχείο επί της ουσίας. Γι' αυτό τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναθεωρηθούν με νομοθετική πρόταση που θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη συνεργασία μεταξύ της ε, του Ευρωπαϊκού Συστήματο Κεντρικών Τραπεζών και του ESS. Καλώ ορίζουμε ιδιαίτερα το γεγονό ότι το σχέδιο έκθεση ε, εξασφαλίζει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων στο θέμα των ε, ε, ισολογισμών, των πληρωμών, των επενδύσεων, ζητώντα γνωμοδοτήσει για τα θέματα αυτά. Είναι επίση απαραίτητο η ΕΚΤ να συμπεριλάβει στο τελικό νομικό κείμενο μια τελογική σκέψη ότι θα γίνει διαβούλευση με την έκθεση για τις νομοθετικές πράξεις που θα εγκριθούν. Είτε είναι πράξη κατεξουσιοδότησης είτε όχι σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για το συζύγιο Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά. Και είμαστε φυσικά πρόθυμοι να βοηθήσουμε στα πιο δύσκολα σημεία ιδιαίτερω σε ό,τι αφορά τι αεροτοπέ άμεσε επενδύσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή και την ΕΚΣ. Και τώρα η συζήτηση έχει πάλι το λόγο. Να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Μόσκα για την γενική της στήριξη και για τα καλά της λόγια. Να ευχαριστήσω επίσης και για το ενδιαφέρον και τη στήριξη των προτάσεων της έκθεσής μου από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eurostat και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα έρθω πάλι σε επαφή μαζί σας έτσι ώστε να έχω περισσότερες λεπτομέρειες από πλευρά σας. Τα θέματα αυτά δεν είναι θρησκευτικής φύσεως, πρέπει να είναι λειτουργικές οι προτάσεις αυτές. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι το κοινό έχει δικαίωμα να λαμβάνει δεδομένα, να έχει στη διάθεσή του δεδομένα υψηλού επίπεδου που να του δίνουν πραγματικές απαντήσεις για το FDI. Πάντα και σαν φοιτητή οικονομικών μου έκανε εντύπωση που το Λουξεμβούργο είναι μία από τις κεντρικές χώρες άμεσων ξένων επενδύσεων. Δεν με πειράζει αυτό. Απλά έχω αμφιβολίες ε, για το αν πράγματι τα χρήματα χρησιμοποιούνται στο Λουξεμβούργο. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί εγώ δεν θέλω απλά να υπάρξουν κάποιες απλές προσαρμογές. Οι διεθνείς οργανισμοί ε, ήδη απασχολούνται με τα θέματα αυτά και κάθε πρόταση από όλα τα θεσμικά όργανα είναι καλοδεχούμενη και νομίζω ότι με τους σκιώδεις θα βρούμε σωστές λύσεις έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια έκθεση που θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε γρήγορα διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Στα πλαίσια της προηγούμενης εντολής υπήρχε μια, ένα ειδικό ενδιαφέρον από το Προεδρείο να ασχοληθεί με τον ε, τριμερή αυτή διάλογο και από ό,τι βλέπω θα διασκεδάσετε με τα θέματα αυτά στο μέλλον αν και δεν υπάρχει και τεράστιο ενδιαφέρον από τα μέλη της Επιτροπής μας. Αυτά. Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε την καλή μέχρι τώρα συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, κύριε Συγητά, ευχαριστώ τους ομιλητές. Στις 12 θα ψηφίσουμε ακριβώς για το δεύτερο τη δεύτερη ανάγνωση του νομοθετήματος για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρημάτων που λαμβάνει υπόψη στην έκθεση Γίγκο και προσβλέπω στον τριγωνικό διάλογο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να οριστικοποιήσουμε σε αυτό το νομοθέτημα. Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται είναι προθεσμία για τις τροπολογίες 19 Μαΐου, εξέταση τροπολογιών 15 ή 16 Ιουνίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή αμέσως μετά την, ε, στην ίδια συνεδρίασή μας και μετά έχει ο Θεός. Θα ακολουθήσει κατά ο τριγωνικός διάλογος και μετά θα θεσπίσουμε το περαιτέρω χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ και τώρα κλείσαμε την πρωινή μας συνεδρίαση και θα έχουμε στις 12 μια κοινή συνεδρίαση με την Λίμπε εδώ στην ίδια αίθουσα για να ψηφίσουμε και να εγκρίνουμε την τελική θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση για τη δέσμη μέτρων κατά του ξεπλήματος χρημάτων. Θα είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό και από πολιτική άποψη. Διακόπτουμε έως τις 12. 12 θα είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ πολύ.